Μία μικρή ανακοίνωση. Πολύ σύντομη. Και θα τα πω στα πολωνικά. Η διάσκεψη των Προέδρων ομόφωνα ενέκρινε την απόφαση για το βραβείο Ζαχάροφ. Πολύ σημαντικό βραβείο, πολύ σημαντική απόφαση. Πέντε εκπρόσωποι της Αραβικής Άνοιξης ε, θα είναι οι άνθρωποι στους οποίους θα απονεμηθεί και θα σας αναγνώσω τα ονόματά τους. Έρτνιε, Μοχαμέτ Μποβαζίζη Στουνέζη. Ασμά Μαχφόους Αιγύπτου. Αχμετ Αλ zubair Αχμετ Αλ Σανούσι, z Λιβύη. Ράζαν Ζεϊτόνε ή Άλλη Φάρτσατ Σύρι. Από τη Συρία. Οι δύο τελευταίοι. Μποαζίζει την Ισία, Μαχμούς Αίγυπτος, Αχμές Αλσανούζη Λιβύη κτλ. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό δείχνουμε την υποστήριξή μας για τα όσα γίνονται στις ε, γειτονικέ αυτές ε, χώρες και δείχνουμε ότι ε, υπάρχει αλληλεγγύη προς τον αραβικό κόσμο προωθούνται οι θεμελιώδεις αξίες μας. Πραγματικά θαυμάζουμε και βραβεύουμε όλους όσους αγωνίζονται στη γειτονική Ήπειρο.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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή αυτού του κοινοβουλίου στην καταστροφική βροχή που έπεσε απόψε το βράδυ στην Τυραλία, Λιγορία και το Σκάνι. Ε, άτομα, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ε, υπάρχουν εκτοδάδε εκτοπισμένοι, σπίτια καταστράφηκαν, χωριά εξαφανίστηκαν εντελώς. Ε, θέλω να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να εκφράσει την αλληλεγγύη του για αυτέ τι περιοχές που καταστράφηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σημειώνουμε την παρατηρήσή σας και περνούμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία επί της αιτήσιας εκθέσεως ε, του Δημοσιολαβητή για το 2010. Ε, ε, μία ψήφους υπέρ, κατά, αποχές.